Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une place. Καλησπέρα. Ελπίζω να βρήκατε θέση να καθίσετε, λέει ο πρόεδρος αστειευόμενος. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει. Ανακοίνωση του συνεδέρφου Γκέγερ σχετικά με πρόταση κανονισμού, με ρύθμιση που έχει σαν στόχο τροποποίηση κανονισμών των διαφόρων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κύριε Γκέγερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εδώ μια πρόταση της Κομισιόν για την υπηρεσία που ασχολείται με τις ε, κεφαλαιαγορές για να προωθήσει την ένωση των κεφαλαίων και έτσι έχουμε περισσότερους άμεσους ελέγχους ε, που αποδίδονται ως αρμοδιότητες της τρεις υπηρεσίες, ειδικότερα στην ΕΣΜΕ. Υπάρχει επίσης μια επανεξέταση του μοντέλου χρηματοδότησης και διακυβέρνησης ε, των ε, υπηρεσιών αυτών, όπως είχε ζητήσει και η δική μας η Επιτροπή. Βεβαίως, μαζί με τις αυξημένες αρμοδιότητες λαμβάνουν και αυξημένους πόρους και εκεί πέρα πρέπει να δούμε για το εάν έχει γίνει ο αναλογός σχεδιασμός όσον αφορά τις ανάγκες τους. Μέχρι στιγμή το μοντέλο χρηματοδότησης ε, των υπηρεσιών λειτουργεί ως εξής 40% του κόστους ε, το φέρει ο κοινοτικός και 60% οι εθνικές εποπτικές αρχές. τα ποσοστά των εθνικών αρχών ε, υπολογίζονται με βάση και τις ψήφους των κρατών στο Σύμβουλιο κάτι το οποίο δεν θεωρώ πολύ δίκαιο πρέπει να σας πω γιατί έχουμε μεγάλες χώρες ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Πολωνία, Ρουμανία που λόγω και του μεγάλου πληθυσμού έχουν ε, πολλές ψήφους στο Συμβούλιο, αλλά λόγω του ιστορικού παρελθόντος έχουν πολύ ασθενή χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ έχουμε ε, χώρες όπως ε, η Γαλλία, η Γερμανία και μια χώρα που ε, δεν θέλω να την ονομάσω, αλλά έχει πολύ μικρό πληθυσμό και μεγάλο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τότε δεν θα πρέπει ο πληθυσμός να αποτελέσει το μέτρο, αλλά η ισχύ του χρηματοπιστωτικού τομέα της κάθε χώρας. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο αυτό. Ειδικά καθώς αυτό είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε έλλειψη πόρων για να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους οι υπηρεσίες αυτές. Βεβαίω. Ε, όπως αντιλαμβάνεστε το Συμβούλιο έχει πολλέ αντιρρήσει, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έχει επιφυλάξει για το εάν ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως ε, κατόπιν ακολούθησε η δική μας αίτηση μιας δικής μας νομικής γνωμοδότησης για να μπορούμε να αντιπαρατάξουμε κάτι στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου το πώς θα ρυθμιστούν τα τέλη θα το καθορίσει τελικά μια πράξη ή κάτι εξουσιοδότηση. Και εδώ πέρα θέλουμε να διασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καθόλου. Οπότε, η δική μου πρόταση είναι πως ε, το κομμάτι της χρηματοδότησης των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει κατά 50% τουλάχιστον να είναι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτός κάπως ακαθόριστος αριθμός οφείλεται στο ότι θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε βάση στο εξής. Εκεί όπου η αποστολή τους είναι ε, καθαρά τεχνικής φύσης, ε, ενίκεια, πληροφορική, ασφάλεια κτλ. Δεν θα πρέπει να καλύπτεται από συνεισφορές ε, των κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων. Με αυτόν τον τρόπο προστατευόμαστε από το ότι μπορεί να προκύψουν ξαφνικά ε, κάποιες ε, ανάγκες, ε, υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες μετά θα εξαρτώνται από άλλους χρηματοδότες και έτσι ίσως υπάρξει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στη μεικτή χρηματοδότηση και άρα τουλάχιστον το διοικητικό κόστος να μπορεί να καλύπτεται στο εκτελεστικό συμβούλιο θέλουμε να υπάρχει η αρχή της ε, απλής ε, πλειοψηφίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής θα περιορίζεται κάπως ε, στο έργο του. Και βεβαίως θα πρέπει ακριβώς υπάρχει προσοχή στην κατάρτιση του shortlist ε, λαμβάνοντα υπόψη και την ισορροπία των φύλων. Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή μας είναι η εκπρόσωπηση του Κοινοβουλίου στο Εκθελεστικό Συμβούλιο. Αυτό το έχουμε προτείνει και σε πολλές άλλες υπηρεσίες ακριβώς για να υπάρχει και πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και μια δημοκρατική λογοδοσία των υπηρεσιών αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέγερ για την παρουσίασή σας η οποία θα μας επιτρέψει έτσι να αντιδράσουμε στις ε, προτάσεις σας. Ποιος θέλει το λόγο? Ο κύριος Σαλβόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, του κύριο Γκάγερ, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, συμφωνώ σε επιτοπλίστων με την θέση της γνωμοδότησης αυτής. Και κυρίως με την γενίκευση των δημοσιονομικών κανονισμών να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Έτσι, Μπορεί να βελτιωθεί η συνοχή, η αποτελεσματικότητα, αλλά και η λογοδοσία των οργανισμών αυτών. Και να βελτιωθεί και η κυβέρνησή τους βέβαια. Τώρα μετά από την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, κύριε Γκάγερ, νομίζω ότι θα ήταν καλό να τονίσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο του προπολογισμού βάση επιδόσεων να δούμε επίσης ποιες είναι, είναι οι συσχετισμοί μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και ποιες οι σχέσεις με τις εθνικές αρχές. Πρέπει να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι όλοι οι οργανισμοί δουλεύουν με όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να αποσφέρουν μια πραγματική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Η δεύτερη, το δεύτερο πράγμα που με απασχολεί είναι το ατέλει. Με τίποτα τα τέλη δεν θα πρέπει να πληρώνονται ε, απευθείας από τις αρχές, γιατί αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα. Και ούτε θα πρέπει να κινδυνεύει η ακαιρεότητα και η ανεξαρτησία των ε, αρχών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Άλλος κανείς. Ο κύριος Άλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάιερ για το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο ε, προτείνει διάφορους κανονισμούς για τις ε, τρεις υπηρεσίες που αφορούν τις χρηματαγορές. Είμαστε πεπισμένοι πως ε, η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ενώ συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση των χρηματαγορών ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Άρα χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες και ισχυρή εποπτεία. Επ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο κλειδί οι αρχές αυτές έτσι ώστε να έχουμε χρηματαγορές με στη βαρύ ρύθμιση για τις τρεις υπηρεσίες, ε, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, την ΕΙΟΠΑ και την ΕΣΜΑ. Συμφωνούμε με την προσέγγιση της Κομισιόν. Η πρόταση της έχει στόχο να δώσει καλύτερες ευκαιρίες για την εποπτεία της αγοράς σε πολλές πτυχές. Ε, την ενίσχυση και την βελτίωση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, την ε, δημιουργία πιο αποτελεσματικού μηχανισμού διακυβέρνησης ε, για να μπορούν οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν αποδοτικά. Θα χρειαστούν επιπλέον θέσεις ε, και πόρους σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν. Για να περάσουμε στην πλευρά των εσόδων, συμφωνούμε με την άποψη του εισηγητή ότι όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση των εποπτικών αρχών πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή θα πρέπει να ανταποκρίνεται το ποσό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στο μέγεθός του για να είναι πιο δίκαιο και πλέον θα πρέπει να υπάρχει και αυξημένος δημοκρατικός έλεγχος μέσω της συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Κύριε Γκαγιέρ, εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των ε, αρχών αυτών, είναι σαν να πρόκειται για μια φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και δεν θα έπρεπε αυτό να θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των εποπτικών αυτών αρχών. Μπορεί να είναι κάτι που θα αποτελέσει επιπλέον πόρους ώστε να μην χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτή είναι η παρατήρηση που θα είχα να κάνω σε αυτά που μας είπατε. Κύριε Γκάιερ, θα ολοκληρώσετε. Ναι, βεβαίως. Να απαντήσω στην ερώτησή σας πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Προς το παρόν, έχω τη στήριξη των ε, συναδέρφων με τους οποίους είχαμε πολύ καλή ε, συνεργασία. Μπορούμε να βρούμε ένα συμφασμό για αυτά που είπε ο κύριος Έλλη αλλά για αυτό που είπατε εσείς, Πρόεδρε, υπάρχει κάτι σημαντικό από το παρελθόν. Και αυτό είναι ότι προσπαθούσαμε πάντα να φροντίσουμε η αρχές αυτές να αποτελούν ε, τη δύναμη ακριβώς των ε, πελατών τους. Συνεπώς, αυτή η συμμετοχή από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ήταν ε, πάρα πολύ περιορισμένη. Είναι, υπάρχουν άλλες αρχές ας πούμε που πιστοποιούν τα αεροπλάνα. Και είναι αλλιώ τα πράγματα όταν έχουμε να κάνουμε με άλλες αρχές. Στην περίπτωση αυτών των τριών πάντως ε, αρχών είναι πολύ σημαντικές για τις υπηρεσίες και μας επιτρέπουν να ε, συνεισφέρουμε σημαντικά στην πιστοποίηση γιατί υποφέρει η αγορά αυτή στην Ευρώπη. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ανεξαρτησίας των αρχών αυτών, η οποία όντως δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι αρχές αυτές να εξαρτώνται πλήρως απόλυτα από την εθνική χρηματοδιώτηση, είτε πρόκειται για την αεροναυτιλία, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Μια που θέλουμε έτσι κι αλλιώ να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των επαπτικών αρχών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι ακριβώς το θέμα αφορά το ποσοστό το οποίο δεν πρέπει να πληρώνουν τόσο η... ο κλάδος αλλά οι εθνικές εποπτικές αρχές και αυτό οδηγεί σε κάποιες αλλαγές ε, της ισορροπής χωρίς να αλλάζει βεβαίως τον χαρακτήρα μιας αφορολογήσης και να μην επηρεάζει την ανεξαρτησία βεβαίως. Ε, δεν είναι συστηματικό θα έλεγα, αλλά εάν ε, πρόκειτο για μια φορολόγηση νομίζω ότι θα ήταν μια απόφαση του Κοινοβουλίου την οποία έχει υποστηρίξει η ομάδα μου και άλλες οπότε εγώ δεν θα είχα και κανένα πρόβλημα. Μα δεν θέλουμε να πληγεί ανεξαρτησία τους. Εννοείται ότι θέλουμε να είναι απόλυτα ανεξάρτητες. Αν όμως το επίπεδο συνεισφοράς καθοριστεί με νομοθετική πράξη, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους οργανισμούς και τις αρχές τις οποίες εποπτεύει η αρχή όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Διακυβέρνησης. Μήπως εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην τηρείται η αρχή ε, διάκρισης των εξουσιών. Αυτό είναι το... Αυτό είναι η απορία μου. Γκάιερ. Ε, ας πω την αλήθεια κυρία Τουή, εμένα δεν με ανισχύει το θέμα. Ίσως είναι και ζήτημα πολιτικής ε, κουλτούρας ε, μεταξύ ημών και μου που δεν συμφωνούμε ίσως 100%. Δηλαδή εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή νομοθετεί για το πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών δεν χρειάζεται να τα αφήνει μετά στην μοίρα τους αλλά να βλέπουμε μετά το πώς εκπληρώνει στην πράξη τις αρμοδιότητες αυτές, ποια προβλήματα συναντάει πια προβλήματα υπάρχουν πιθανώς και με την ομοθεσία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που αποφασίζουμε κάτι με τις καλύτερες των προθέσεων και μετά αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή. Όλα αυτά θα τα λαμβάνουμε ως πληροφορία πολύ πιο άμεσα αν υπάρχει ένας εκπρόσωπος, μία εκπρόσωπος ε, του Κοινοβουλίου στην καθημερινή λειτουργία του κάθε οργανισμού. Θεωρώ ότι αυτό θα μας κάθισε πιο εξοικειωμένους με την καθημερινή λειτουργία αυτών των οργανισμών από το να δίνουμε μόνο κάποιες γενικές κατευθύνσεις ε, και να καθορίζουμε το νομικό πλαίσιο και μετά να ελπίζουμε ότι θα συμβεί το καλύτερο. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Μπορεί βεβαίω. Κάποιο να έχει άλλη άποψη και να απορρίψει, να την πρότασή μου. Καλώς. Σε αυτό θα σταματήσουμε. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 την 5η 21 του μηνός και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 10 Ιουλίου. Κύριε Γκέγερ, Είστε πάντα εισηγητής. Πρόκειται για άλλη γνωμοδότηση, για πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πριν υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησής του βασικά, για να ξέρουμε ποια είναι η θέση των ομάδων στην υπόθεση αυτή που έχει σαν θέμα τη νέα ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διάφορα ταμεία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικό Ταμείο, Συνοχής, Γεωργικό και Ανάπτυξης της Υπέθρου, ε, το Ταμείο για την Αλία και τη Θάλασσα. Όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν καλύπτονται από μια ρύθμιση και ο κύριος Γκάγερ θέλει να ξέρει την άποψη των σχεδόν εισηγητών για την τροποποίηση αυτή. Έχετε το λόγο κύριε Γκάγερ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Πράγματι μοιάζει πολύ τεχνικός ο τίτλος, αλλά πίσω από αυτό υποκρίνεται ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι συνδιαπραγματεύτηκαν το πλαίσιο οδηγίας θα θυμούνται πως η πρόταση της Κομισιόν πήγαινε να υπάρξει, στην κατεύθυνση να υπάρξει ένα αποθεματικό απόδοσης ε, στο Ταμείο Συνοχής το οποίο θα απελευθερωνόταν όταν και αν τα κράτη ή οι περιφέρειες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων ε, πληρώσαν ορισμένους όρους. Αυτό τότε είχε ερμηνευτεί ως ε, ένα κρυφό μέτρο λιτότητας, ε, το οποίο πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο και σε κάποιους άλλους ε, φάνηκε ως ένα έργο ελέγχου της απόδοσης. Ε, τώρα η Κομισιόν θέλει να μην ενισχύει πλέον το απόθεμα αυτό επιχειρησιακά προγράμματα όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έτσι βεβαίως ε, θα έχουμε φτάσει στο εξής. Αυτό το οποίο φοβόμασταν πριν από χρόνια. Δηλαδή έχουμε ένα μέσο λιτότητας το οποίο υλοποιήθηκε για τα λεφτά αυτά πλέον δεν είναι στην διάθεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είχε διατεθεί για κάτι στο οποίο είχαν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη, αλλά μετά δεν πηγαίνει σε κοινή διαχείριση των κρατών μελών, αλλά σε απευθείας διαχείριση της Κομισιόν. Κάτι το οποίο δεν αφαιρεί μόνο λεφτά από τα υπηρεσιακά προγράμματα, αλλά αφαιρεί και την ε, συνδιαχείριση των κρατών μελών, γιατί είναι υπό την άμεση διαχείριση της Κομισιόν. και αυτό αιτιολογήθηκε από την Κομισιόν ως προάγγελος του επόμενου ΠΔΠ που εγώ είπα καθίστε ρε παιδιά να το διαπραγματευτούμε πρώτα και να μπορέσουμε να κρίνουμε εάν λειτουργήσει κάτι τέτοιο ή όχι. Και τέλος η Κομισιόν εξετάζει τακτικά την τήρηση των επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων και αυτό τελευταία φορά, η επόμενη φορά θα γίνει τέλος του 19. Τέλος ε, του 2019. Έχουμε δηλαδή ε, ένα χρόνο μέχρι να τεθεί ενισχύει το νέο πιδελταπή. Γιατί ε, το να το πούμε αυτό πιλωτική προσπάθεια για να δούμε αν μπορεί να γίνει στην πράξη κάτι τέτοιο μου φαίνεται κάπως ε, περίεργη η αιτιολόγηση. Εμείς ε, μέχρι τώρα λέγαμε ότι εκεί όπου υπάρχουν νέες αρμοδιότητες θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει και φρέσκο χρήμα και από το Ταμείο Συνοχής. Όλες αυτές οι σκέψεις με οδηγούν και εδώ πέρα συμφωνώ με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και στην Επιτροπή Περιφερειακής ε, Πολιτικής ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την ε, πρόταση της Κομισιόν. Προτείνω λοιπόν να απορρίψουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Γαγιέρ. Η σκιώδες εισηγητές τώρα. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα των χωρών μελών, για την ανάπτυξη, την οικονομική, για την απασχόληση, για τις αλλαγές που γίνονται καθημερινά στον κόσμο. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην μπερδεύουμε τα θέματα μεταξύ τους. Είναι αλήθεια ότι η πολιτική συνοχής βοηθάει για να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε μια χώρα μέλος, ναι. Αλλά αν θέλουμε ένα, ένα πρόγραμμα για τις διαφορετικές αλλαγές, αν αλλάζουμε τους κανόνες, αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Το αποθεματικό της ε, απόδοσης, performance ε, reserve, είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού που έκαναν οι χώρες μέλη. Το αποθεματικό αυτό πρέπει να διατηρείται για τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Είναι και θέμα προβλεψιμότητας για τους δικαιούχους των ε, Ταμείων Συνοχής, των κονδυλίων. Καταλαβαίνω τη θέση του εισηγητή βέβαια και ακούω διάφορα και από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχω πάντως κάποια αμφιβολία για αυτό το θέμα. Και τι σημαίνει αυτό για την ελαστικότητα. Δηλαδή, αν δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες μέλη σε θελοντική βάση να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν σε αυτή την περίφημη performance reserve, αν τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, μήπως πρέπει να απορρίψουμε την ευελιξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι διαφορετικές αλλαγές, ακόμα και στο νέο πρόγραμμα, θα γίνουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο αλλά και σε εθελοντική βάση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα κονδύλια για αυτούς τους στόχους. Και κάτι άλλο που με ενοχλεί. Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δαπάνες που θα έπρεπε να αναλάβει ο εθνικός προϋπολογισμός τρέχουσες δαπάνες δηλαδή, ε, δαπάνες λειτουργίας. Όλα αυτά πρέπει να καλύπτονται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Οι μεταρρυθμίσεις επίσης πρέπει να στηρίζονται σε ένα βαθμό και από τον εθνικό προϋπολογισμό. Αν υπάρχει βέβαια κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα, εντάξει. Αλλά να παίρνουμε χρήματα από την πολιτική συνοχής, ακόμα και αν είναι από την ε, performance reserve, δεν είναι σωστό. Όλα αυτά που λέω δείχνουν ότι είμαι κάπως μοιρασμένο. Εξαιτίας αυτής της εθελοντικής βάσης και της ευελιξίας. Αν εμείς μπορούμε να πούμε, όχι, ακόμα και αν το κράτος μέλος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το παθηματικό, εμείς είμαστε κατά, δεν θα τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν ξέρω, έχω τις αμφιβολίες μου. Ελπίζω με τη συζήτηση να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάπως καλύτερα τι τελικά πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουρμέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ για τα καλά του λόγια, για τα απλά του λόγια που κατέστησαν νομίζω σαφές ε, το πόσο δύσκολο είναι αυτό το πακέτο το οποίο συζητάμε και δεν είμαι τόσο σίγουρος για ναι, το αν είναι τόσο καλή ιδέα να τα συζητάμε όλα υπό έναν τίτλο. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πτυχές ε, της υπόθεσης αυτής ε, αφενός ε, αυτή, την οποία πάντα υπενθυμίζουν τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να απλοποιήσουν τα πράγματα δηλαδή Ε, δεν αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας εδώ πέρα. Από την άλλη πρέπει να είμαστε σαφείς όταν έχουμε τόσα πολλά είδη επιδοτήσεων ε, υπό έναν τίτλο θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές γιατί βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε μία έννοια αντιμετώπιση στα πάντα και επιπλέον νομίζω θα πρέπει ε, να δούμε και τι μπορούμε τελικά να πληρώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και έχουμε ε, δημιουργήσει τόσες πολλές προσδοκίες που αναγκαστικά θα υπάρξουν απογοητεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το τι μπορούμε να απλοποιήσουμε. Απλοποίηση σημαίνει και διαφάνεια. Και θα πρέπει ακριβώς ε, να δούμε και την ε, ουσία. Και να κάνουμε λίγα πράγματα και να τα κάνουμε σωστά. Και ε, αλλιώς θα έχουν χάσει και την εικόνα οι πολίτες και θα έχουμε και προγράμματα που δεν θα χρησιμοποιούνται και δεν θα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει ακριβώς να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, τον γόρδιο δεσμό αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις αυτή τη στιγμή. Οπότε συνάδελφοι, αν θέλετε να πάρετε το λόγο μπορείτε. Όχι. Ωραία, τότε θα ζητήσω από τον κύριο Γκάγερα να κλείσει. Δεν χρειάζεται. Μου κάνει νόημα πως δεν θέλει. Να σας πω ότι το σχέδιο έκθεσης θα σας υποβληθεί στη συνεδρίαση της 9ης ή 10ης Ιουλίου και ότι στις 12 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ότι θα αποφασίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού στο 29-30 Αυγούστου και 21 Νοεμβρίου η Ρέτζη, που είναι αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή, θα αποφασίσει και εκείνη. Τώρα, θα ακούσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε δύο σημαντικές αποστολές, τη μία στη Μολδαβία και την άλλη στην Ισπανία. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας που πήγε στην ε, Μολδαβία, τον Ζίκφριτ Μουριζάν, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης ε, για την αποστολή αυτή. Και έπειτα οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή, την, ε, ο κ. Φερνάντες, η κ. Γουάρδια Ζαμπάλ, και ο κ. Φόντου θα μπορέσουν να μας κάνουν τη δική τους παρουσίαση αν θέλουν να μας δώσουν την αίσθηση που αποκόμισαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, επισκεφθήκαμε τη Δημοκρατία της Μολδαβία ε, μεταξύ της 1ης και της 6ης Μαΐου για μια εντατική και μακρά επίσκεψη. Ξεκινήσαμε λοιπόν ε, την ε, Δευτέρα με, είχαμε 23 συνεδριάσεις με την ADF Γαρτιτσαμπάλ, τον κύριο Κόλμελ και τον κύριο Φερνάντες βασικός στόχος ήταν να αξιολογήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην Ένωση και την Μολδαβία και ιδιαίτερα την ε, οικονομική σχέση μας και την ε, δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα αυτή. Η, Μολδαβία έχει, η Μολδόβα έχει ε, συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση έχει ξεκινήσει δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό μονοπάτι. Τι κάναμε λοιπόν στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Είχαμε ε, συνεδριάσεις, ε, επαφές υψηλού πολιτικού επίπεδου μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ήταν εκεί και μια αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ και είχαμε πολιτικής φύσης συνεδριάσεις με τους συναδέλφους της ΑΦΕΤ και στη συνέχεια είχαμε χωριστέ συνεδριάσεις στον τομέα του προπολογισμού και επισκεφθήκαμε πολλά project που χρηματοδοτώνται από κονδυλία της Ένωσης. Συναντήσαμε τον πρόεδρο της χώρας, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, συναντήσαμε ε, βουλευτές ε, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, είχαμε και επαφές με ε, την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση, είχαμε επαφές με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Είχαμε, ε, πιστεύω πως αποκομίσαμε μια καλή εικόνα για την κατάσταση της χώρας και για την ε, δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βεβαίω ε, λεπτομέρειες θα δείτε στην έκθεση της Επιτροπής μας, αλλά να σας πω ποια ήταν τα βασικά μας πορίσματα. Πρόκειται για μια χώρα που έχει μπει στο δρόμο της Ευρώπης μια χώρα όπου και εμείς, εμείς συμμετέχουμε πολύ. Μάλλον είμαστε εντόνως αναμεμειγμένοι πολιτικά. Γείται μια κυβέρνηση που σχηματίστηκε επί τη βάση μιας ad πλειοψηφίας που δεν προέκυψε όμως ως πλειοψηφία μετά τις τελευταίες εκλογές. Μετά τις τελευταίες εκλογές υπήρχε μια υπερευρωπαϊκή πλειοψηφία αλλά το κύριο κόμμα μέσω διαφόρων ε, προσχωρήσεων μπόρεσε να αποκτήσει περισσότερα μέλη στο Κοινοβούλιο που προέρχονται από, διάφορες, ε, όμως, από διάφορα κόμματα και να επηρεάσει και την τοπική ε, διακυβέρνηση. Να σας πω κάποια στοιχεία. Το Κοινοβούλιο είχε 220 δημάρχους ενώ τώρα έχουν 680 οι δημάρχους από το 900, η κυβέρνηση δηλαδή. Πολιτικός ε, ένα σημείο είναι πολύ σημαντικό και το... Αυτό είναι η κυβέρνηση. Έχουμε τη συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδόβα και ε, το κόμμα αυτό ε, που κυβερνά παρουσιάζεται ως υπερευρωπαϊκό, αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η εφαρμογή. Δικό μας συμπέρασμα, το οποίο ε, συμφωνούν και οι συνάδελφοι της ΑΦΕΤ, είναι ότι η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης είναι πολύ βασική. Αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, όχι μόνο η οθέτηση μιας νομοθεσίας για να δημιουργηθεί ένας θεσμός, ας πούμε, ή ο οργανισμός κατά της διαφθοράς ή υπέρ της και θεσμοί που είναι πολύ σημαντικοί για μας γιατί εξασφαλίζουν ε, ότι οι δικαιούχοι των ευρωπαϊκών κονδυλίων φτάνουν, παίρνουν τα χρήματα που δικαιούνται ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στελεχώνονται σωστά. Η χώρα θέλει να προχωρήσει προς την Ευρώπη, αλλά αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι ο κόσμος γνωρίζει τα πλονεκτήματα της στενότερης ε, επαφής με την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της χώρας είναι φιλορώσος και διαρκώς μιλάει για τα ωφέλη της συνεργασίας με την ε, Ρωσία και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα ωφέλη του, της περισσότερης επαφής με την Ένωση. Εμείς πρέπει αυτό να το ε, αντιμετωπίσουμε μέσω της αντιπροσωπείας μας εκεί, μέσω των επισκέψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να μιλήσουμε για τα ωφέλη της στενότερης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ ισχυροί και τα μηνύματά μας να είναι πολύ έντονα για το κράτος δικαίου, την εξαρτησία του δικαστικού σώματος, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, το ξέπλυμα χρήματος και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι το μίσο που πρέπει να είμαστε πολύ στεναροί. Και φυσικά αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο θα πανώνται τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά επιτόπου. Τώρα λοιπόν έχουμε δύο ακόμα στοιχεία που θα ήθελα να δούμε. Καταρχά, πέρσι είπαμε στην Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν για τη χορήγηση ε, ε, χρημάτων υπό αυστηρούς όρους και είπαμε ότι από τη στιγμή που θα πληρώνται οι όροι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την αποδέσμευση αυτών των χρημάτων από την Κομισιόν αλλά όχι πριν την πλήρωση των όρων που συνδέονται στενά με το κράτος δικαίου, την αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση, τόσο πιο σύντομα θα πάρουμε και τα χρήματα. Τελευταία μου ιδέα, Πρόεδρε, αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα ευρωπαϊκά project. Επισκεφθήκαμε σχολεία που είχαν τελείως ανακαινιστεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλου είδους εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά χρήματα. Επισκεφθήκαμε νοσοκομεία που έχουν ανακαινιστεί με τα ευρωπαϊκά χρήματα, ε, δρόμους που έχουν φτιαχτεί ε, επίσης, ε, συστήματα θέρμανσης που είναι περιβαλλοντικά ε, φιλικά προς το περιβάλλον και έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά χρήματα για τα σχόλια. Από όσο μπορούσαμε να κρίνουμε τα ωφέλη των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι συγκεκριμένα και όντως εξυπηρετούν τον κόσμο. Απλά θέλουμε ο κόσμος να ξέρει ότι προέρχονται από την Ένωση. για οι φιλορώσοι λένε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο υποσχέσεις ε, και λόγια, αλλά δεν κάνουν τίποτα συγκεκριμένο. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε στη χώρα υπό όρους να ζηταπετούμε μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένες. Και τα project που είδαμε πιστεύω πως με λίγα χρήματα, μικρά ποσά μπορούν να γίνουν πολλά θετικά για τον κόσμο της χώρας αυτής στην ανατολική μας γειτονιά. Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ ε, για αυτή σας την αναφορά. Ίσως θέλετε κυρία Κουαρτιαθαμπάλ να συμπληρώσετε κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια μόνο, γιατί πιστεύω πως ο κύριος Μουρεσάν έκανε μια τέλεια ανάλυση για την αποστολή μας και τις ε, συνεδριάσεις και τις επαφές που είχαμε. Κάτι ακόμα, ένα περιστατικό, γιατί το πρώτο τμήμα το μοιραστήκαμε με την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων και Έχουμε πολύ διαφορετικό τρόπο να, βλέπουμε την ε, αποστολή. Για όσους δεν, γνωρίζονται, ήταν πολύ δεν γνωρίζουν την Μολδάβα, ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρώτο τμήμα για να καταλάβουμε ε, τις σχέσεις ανάμεσα στη χώρα αυτή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν κάπως πολύ γενικά όλα αυτά για μια αποστολή του προϋπολογισμού και ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον το δεύτερο κομμάτι, όπου μπορέσαμε να μιλήσουμε για χρήματα, για οικονομική βοήθεια, για project συγκεκριμένα που άμεσα χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Είναι καλό δηλαδή να γίνονται κοινέ αποστολές, όμως κάποιες φορές οι στόχοι είναι πολύ διαφορετικοί και νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο χάνουμε λίγο χρόνο. Ήταν ενδιαφέρον το πρώτο τμήμα, όμως νομίζω πως ε, ε, δεν έχουμε κοινή οπτική. Και έπειτα, για να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. στο τέλος, πρέπει να γίνει μια πολιτική εξήγηση και επικοινωνίας πολύ καλύτερη όσον αφορά τα ωφέλη των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από την βοήθεια τη χρηματοδοτική που είναι άμεση, όλα τα μέσα, τα συμπληρωματικά όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την εξωτερική εντολή της ΜΠΕΙ, το νέο σχέδιο, επενδυτικό σχέδιο και στην πραγματικότητα δεν ξέραν τι τους λέγαμε, δεν είχαν ιδέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει μια τέτοια πολιτική επικοινωνία ώστε να φτάσουμε περισσότερο και στους θεσμούς, δηλαδή εδώ στην κυβέρνηση, αλλά και στις επιχειρήσεις, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης και στήριξης project. Πρέπει δηλαδή να βελτιώσουμε αυτό το τμήμα της επικοινωνίας. Γιατί δεν συμβαίνει μόνο στη Μολδάβα αυτό βέβαια, συμβαίνει και μέσα στις χώρες της Ένωσης. Πολλές φορές ε, πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας στρατηγική. Κολμέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Ζίγκφριντ Μούρεσαν, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή έκθεση και πραγματικά οργάνωσε πάρα πολύ καλά το ταξίδι, ήταν πάρα πολύ καλό ταξίδι και πρέπει να γίνονται αυτές οι αποστολές για να σκεφτόμαστε το τι γίνεται σε αυτές τις ε, χώρες ε, που είναι υποψήφιες, τι μπορούμε ρεαλιστικά να περιμένουμε και τι όχι. Και βλέπουμε εκεί πέρα ότι υπάρχουν χωριά που δεν έχουν ούτε ίδρυψη ούτε αποχέτευση. Και δεν μπορούμε βεβαίω με όση καλή θέληση και να έχουμε ε, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μιας δεκαετίας ας πούμε, να έχουν τις προδιαγραφές ε, που αναμένουμε από ένα κράτος μέλος. Ε, δεν κατηγορούμε βέβαια τον κόσμο επειδή είναι φτωχός, αλλά ε, ακριβώς βλέπουμε έτσι και στα πεταχτά και τις δυνατότητες της διοίκησης, οι οποίες επίσης χρήζουν κάποιας αναβάθμισης. Οπότε όταν μιλάμε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιες χώρες ε, δεν πρέπει να κινούμαστε και πάρα πολύ γρήγορα. Αλλιώ ε, απαιτούμε και πάρα πολλά από αυτές τις χώρες. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει το λόγο. Στην ουσία, κύριε Μούρισαν, Σιγά, λέμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έναν μηχανισμό πάρα πολύ περίπλοκο που θέλει να αποφύγει βέβαια κάθε κίνδυνο. Όταν όμως βλέπετε τους θεσμούς στη Μολδαβία δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου των ε, δημοσίων ε, οικονομικών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί μόνο αν οι χώρες έχουν τέτοια δυνατότητα θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό λιγότερο περίπλοκο. Οπότε δεν ξέρω, λέτε ότι θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τότε θα έπρεπε να έχει ένα σύστημα ελέγχου των οικονομικών. Είναι αναγκαίο. Ναι, Πρόεδρε, χωρίς καμία αμφιβολία. Ακόμα μένει μακρύς ο δρόμος για την Μολδαβία αν κάποια μέρα γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν αυτό είναι σαφές και σε εκείνους και σε μας ότι η χώρα άλλο παρά έχει καλύψει τα κριτήρια που πρέπει να καλύπτει μια χώρα για να ανταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι μεταρρυθμίσεις. Αυτός θα είναι ο δρόμος για την ένταξη. Όταν αρχίσουμε να μιλάμε για ένταξη και οι άνθρωποι στις δικές μας τις χώρες θα πρέπει να νιώθουν ότι η Μολδαβία είναι έτοιμη να ενταχθεί. Γιατί μόνο τότε θα συστήσουμε στους λαούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών την ένταξη της Μολδαβίας. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια εκεί. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι στηρίζουμε την Μολδαβία στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Και ναι, το θέμα της νομοποίησης παράνομου χρήματος, η εξηγένωση των οικονομικών, ε, χρηστή δημόσια δίκηση, όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις, ναι. Η Όλαφ είναι παρούσα εκεί όταν πρόκειται για απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά πάντως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από χρηστή οικονομική διαχείριση. Η χώρα δεν πρέπει να είναι μέρος κανένας κυκλώματος νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και εμείς έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Βρίσκεται στον ε, σωστό δρόμο παρόλο που ο δρόμος αυτός είναι μακρύς. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μουρισάν, την κυρία Γαζεθαμπάλ και τον κύριο Κολμέλ που μοιράστηκαν μαζί μας τα συμπεράσματα που έβγαλαν από την αποστολή αυτή στην Μολδαβία. Ερχόμαστε τώρα στη χώρα των Βάσκων. Ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, την Ισπανία. Έτσι. Την Παρασκευή πέρασα μια υπέροχη βραδιά ποδοσφαιρική. Λοιπόν, κυρία Καστιαφαμπάλ, σας ακούμε, μια από εσείς προεδρεύσατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, ήταν τιμή για μένα να είμαι πρόεδρος της αντιπροσωπείας αυτής στη δικιά μου περιφέρεια. 7 και 8 Μαΐου έλαβε χώρα. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σε αυτές τις δύο μέρες και η ιδέα ήταν να υποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από αυτές τις δύο μέρες για να μπορέσουμε να δείξουμε στους ευρωβουλευτές μια πραγματική εικόνα του πώς γίνεται η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα των Βάσκων και πώς τα κονδύλια αυτά βοηθούν να υλοποιηθούν πολιτικές και σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η αντιπροσωπή αυτή είχε ένα θεσμικό σκέλος και είναι σημαντικό το ότι μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με τους θεσμούς στη χώρα των Βάσκων, την βασκική κυβέρνηση, ε, τα δημαρχία, για να δούμε και τα διάφορα επίπεδα πώς δηλαδή υλοποιούνται πολιτικές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε μια γενική συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027 με λεπτομέρειες για πολιτικές που να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλον, κατοικία, ε, φροντίδα για τους μετανάστες, απασχόληση, ισότητα. Είδαμε λίγο απ' όλα. Και είδαμε και την αστική ε, μεταρρύθμιση, δηλαδή τι έγινε στο Μπιλμπάο με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς άλλαξε η πόλη. Το δεύτερο σκέλος ήταν επαφή με τις επιχειρήσεις και πώς ε, χρησιμοποιούνται, πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε τι προϊόντα καταλήγουν και σε τι αποτελέσματα γενικά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες συναντηθήκαμε είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα Horizon 2020. Είδαμε μεγάλες επιχειρήσεις αερο ε, για παράδειγμα αλλά και μικρές που με 50.000 ευρώ από το Horizon 2020 κάνουν έρευνα για τον καρκίνο ή μια άλλη φτιάχνει ένα μοντέλο ανανεώσιμης ενέργειας. Είδαμε επίσης το κρατικό πανεπιστήμιο της χώρας των Βάσκων και τα διάφορα τμήματά του πώς κάνουν έρευνα. Και αυτό που είχαμε σχέση με το Horizon 2020. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν μπορώ να είμαι αντικειμενική γιατί βλέπετε είναι δικιά μου η γη, η περιοχή είχα την τύχη να προεδρεύω τις αντιπροσωπείες αυτής, αλλά πιστεύω όμως πραγματικά ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Και οι στόχοι, τους οποίους εγώ έθεσα τουλάχιστον όταν πρότεινα αυτή την αποστολή, υλοποιήθηκαν και θεσμικά και επιχειρηματικά. Είδαμε πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς αποτελούν προστιθέμενη αξία για την έρευνα και την ανάπτυξη. Είδαμε θετικές πρακτικές, θετικά αποτελέσματα. Οπότε ελπίζω τουλάχιστον η αποστολή αυτή να ήταν ικανοποιητική για όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε όλες τις συναντήσεις και ευχαριστώ πολύ τη γραμματεία. Δεν ήταν εύκολο σε δύο μέρες με τόσες επισκέψεις, τόσες επαφές Είχαμε και συνάντηση με διάφορες επιχειρήσεις που σε πέντε λεπτά η καθεμία μας παρουσίασαν τα προϊόντα τους για να μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν ε, δύσκολο το οργανωτικό σκέλος. Πάντως πήγε πολύ καλά πιστεύω. Οπότε ευχαριστώ και τη γραμματεία. Τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκτός μικροφώνου όμως. Ευχαριστούμε που με τέτοια αντικειμενικότητα παρουσιάσατε την ε, επίσκεψη. Οι δυνατότητες που έχει η χώρα των Βάσκων και η καλή χρήση που κάνει των ευρωπαϊκών κονδυλίων ήταν το θέμα. Ωραία, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους άλλους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή, αλλά σας έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Οπότε είσαστε και πρόεδρος αντιπροσωπείας και αυτοί που παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο για αυτήν την ε, αποστολή, προχωράμε στον κύριο Μούρεσάν, ο οποίος θέλω να μας βοηθήσει να δούμε τον, την ε, τροποποιητική ε, ανακοίνωση προπολογισμού αριθμό 3 όσον αφορά τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Πώς θα επεκταθεί η διευκόλυνση αυτή δηλαδή. Παρακαλώ κύριε Μουρισάν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να αναλύσουμε τώρα τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 μέσα στο οποίο η Κομισιόν προτείνει να καταναμηθούν 550 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των προσφύγων στην Τουρκία το 2018. Γνωρίζουμε ακριβώ ε, από που ερχόμαστε. Είχαμε δύο χρόνια αυτού του μέσου. Τρία δισεκατομμύρια. Ένα δισεκατομμύριο από τον κοινωνικό προπολογισμό και δύο από τα κράτη-μέλη. Μετά υπήρξε η πρόταση να δοθεί μια συνέχεια. Εμείς είμαστε υπέρ της παράτασης. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία. Στηρίζει τους πρόσφυγες επιτόπου και δεν κινδυνεύουν να με το να οδεύουν προς την Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς ε, το Κοινοβούλιο στο σύνολό του είναι υπέρ της παράτασης. Ε, εμείς ε, πάντα λέγαμε το εξής. Συμφωνούμε με την παράταση, αλλά θέλουμε να την χρηματοδοτήσουμε όπως χρηματοδοτήσαμε και το πρώτο μέσο. Ένα δισεκατομμύριο από τον προπολογισμό της κοινότητας και δύο από τα κράτη-μέλη. Και είπαμε επίσης ότι θέλουμε νέους πόρους. Γιατί είπαμε ότι οι νέες προτεραιότητες πρέπει να έχουν νέους πόρους ε, και είπαμε ότι το πι δελτα πι ήδη έπρεπε να κάνει τόσο πολλά πράγματα που δεν προβλεπόταν το 2013 όταν αποφασίστηκε. Το ΕΦΣΙ, ΕΦΣΙ2, ΕΦΣΙ για την Αφρική, Ταμείο για την Αφρική, το Μέσο για τους πρόσφυγες, πολλά έργα για τη μετανάστευση. Οπότε είπαμε νέο χρήμα και είπαμε κατά κανέναν τρόπο δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν υφιστάμενα προγράμματα. Αυτό ήταν η απόφαση του Κοινοβουλίου που ελήφθη σε πολλές ε, συνεδριάσεις επιτροπή με τους συντονιστές και με όλους τους βουλευτές τώρα η Κομισιόν πρότεινε την εξή ε, χρηματοδότηση για το μέσο για τους πρόσφυγες στην Τουρκία για το 2018 πρότεινε να δοθούν 505 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 50 από αυτά είναι συγκεκριμένα για ανθρωπιστική βοήθεια και 500 είναι νέοι πόροι. 256 από το περιθώριο στον τίτλο 4 και 243,8 από το συνολικό αποθεματικό των δεσμεύσεων. Οπότε βασικά η Κομισιόν τώρα προτείνει ένα διορθωτικό προϋπολογισμό που προβλέπει 500 εκατομμύρια ευρώ νέων πόρων ε, από τα αποθεματικά. Έτσι δεν διακινδυνεύει κάποιο υφιστάμενο πρόγραμμα και έχουμε και κάποιο περιθώριο για απρόβλεπτα του επομένου έτους. Είπαμε ότι θέλουμε νέα κονδύλια, όχι αναδιατάξεις και το αποθεματικό το οποίο θα μείνει να είναι αρκετό και για αλλά απρόβλεπτα να μην δηλαδή το απορροφήσουμε όλο γιατί δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γίνει ένα σεισμός ή κάτι τέτοιο και τώρα η Κομισιόν προτείνει έναν διορθωτικό προπολογισμό που προβλέπει 500 εκατομμύρια ευρώ σε νέους πόρους δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσο θα είναι ο προπολογισμό του 19 και μπορώ να πω το εξής για το 18 πήραμε αυτό το οποίο θέλαμε και γι' αυτό λέω ότι επί τη βάση αυτού του διορθωτικού προβλησμού δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τον απορρίψουμε. Γι' αυτό η δική μου πρόταση είναι να δεχτούμε αυτόν τον προβλησμό. Αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή οικονομικά. Επίση, πολιτικά είναι σημαντικό να δώσουμε το πράσινο φω στον διορθωτικό προβολισμό, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προβλεψιμότητα για την στήριξη των προσφύγων. Έχουμε επισκεφτεί την Τουρκία, έχουμε επισκεφτεί την Ιορδανία και τον Λίβανο πριν από δύο χρόνια μου και εγώ εκεί και πέρσι την Τινησία και σε όλες αυτές τις αποστολές ήταν πόσο σημαντική είναι η προβλεψιμότητα για να χρηματοδοτήσουμε σχολεία αυτά πρέπει να είναι γνωστά δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο το αργότερο για το αν θα έχουν ε, χρηματοδότηση του χρόνου για να προλάβουν δασκάλους κτλ. Και, και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς για να προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Αλλιώ ε, καταλήγει κανεί ε, θύμα της προπαγάνδας των τρομοκρατικών οργανώσεων. Γι' αυτό ακριβώς και το έχω συζητήσει αυτό με τον Γενικό Εισηγητή του 2019 λέμε ότι τώρα πολιτικά πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως και έχουμε όλα τα επιχειρήματα. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και πήραμε αυτό το οποίο θέλαμε για το 2018. Αλλά πρέπει να τα πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε και για το 2018. Η πρόταση χρηματοδότησης που έχει το Συμβούλιο Επιτάπτωση είναι 2 δισεκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολογισμό και ένα δισεκατομμύριο από τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αν δώσουμε 2 δισεκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολογισμό είτε θα υπάρξουν αναδιατάξεις ε, του χρόνου, δηλαδή επηρεάζονται τα υφιστάμενα έργα ή εάν ε, έχουμε νέους πόρους από το αποθεματικό τότε δεν θα απομείνει τίποτα στο αποθεματικό. Γι' αυτό θα έλεγα όχι στο να πάρουμε 2 δισεκατομμύρια από τον κοινωτικό περιπολισμό και μόνο ένα από τα κράτη-μέλη. Η θέση μας ήταν σαφής. Όπως είπα, 1 δισεκατομμύριο από τον προπολογισμό και 2 από τα κράτη-μέλη. Το 18 πήραμε αυτό το οποίο θέλαμε, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτόν τον προπολογισμό, έτσι θα υπάρχει πρόβλεψιμότητα, σταθερότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις διαπραγματεύσεις του 19 πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, δυνατοί για να υπάρχει μια τελική χρηματοδότηση του μέσου αυτού και τα έχω συζητήσει αυτά και με τον Γενικό Εισηγητή του 2019 εις βάθος και συμφωνούμε σε αυτό ότι δηλαδή πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως στον διορθωτικό προπολογισμό, να παραμείνουμε ενωμένοι και το πράσινο φως που δίνουμε τώρα δεν παδικάζει καθόλου τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως αρχή του προπολογισμού για τον προπολογισμό του 19. Δηλαδή, εάν δεν είναι το μέσο αυτό όπως ε, το θέμε, δεν θα συμφωνήσουμε στην συνδιαλλαγή, αλλά αυτό θα το κρίνουμε αργότερα και βεβαίως δεν μπορούμε να περιμένουμε τη χρηματοδότηση του 18 μέχρι να ολοκληρωθεί η συνδιαλλαγή μέχρι το τέλος του έτους δηλαδή. Γι' αυτό λέω να υπερψηφίσουμε και να είμαστε ενωμένοι για να πάρουμε και το 19 όσα θέλαμε όπως έγινε και το 18. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, εισηγητά κάθε πράγμα στο καιρό του και η συνέχεια φαίνεται ε, ότι είναι προβληματική. Ο κύριος Κόλμελ, ως σκιώδης εισηγητής, ποια είναι η δική σας γνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι θα ευχαριστήσω τον Ζίγφριντ ε, Μουρεσάν ε, ή τα είπε τα ουσιαστικά. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Επιτροπή του Προϋπολογισμού να ζητήσουμε πέρα από τα απαραίτητα κονδύλια να υπάρξει μια πολιτική λύση για το θέμα των προσφύγων. Αλλιώς ε, θεραπεύουμε τα συμπτώματα αλλά όχι την αιτία. Είναι σημαντικό. Αν ε, δεν το έχουμε αυτό κατά νου, συνεχώς θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Δηλαδή, λαμβάνουμε αποφάσεις με τη δικασία του κατεπήγοντος το οποίο μπορεί πράγματι να ισχύει, αλλά η αιτία είναι ότι θα πρέπει να δούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ποια πολιτική ασύλου θέλουμε και όταν ε, πραγματικά συμφωνήσουμε σε αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε σοβαρά ποια λεφτά θα δώσουμε πού. Θεωρώ ότι στον τομέα της διαμονής ε, της ε, Τουρκίας ε, παρέχουμε βοήθεια. Υπάρχουν και άλλες ε, δυνατότητες ε, και αυτή την στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα είναι πιο αποτελεσματικά τα λεφτά μας γιατί δεν έχει γίνει η βασική δουλειά. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να πιέσουμε και να πούμε η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα συμφωνήσει μόνο εάν γίνει και αυτή η σωστή δουλειά. Ευχαριστούμε κύριε Κόλμελ. Κυρία Γιατερμάκη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ ευχαριστώ τον Μούρισαν για την ε, καλή, το καλό σχέδιο που έχει ετοιμάσει. Μπορώ να στηρίξω κι εγώ αυτή την τροποποίηση του προπολογισμού. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν σε αυτό το στάδιο να μην τοποθετηθούμε για τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς, αλλά για τη διαδικασία του 2019. Και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής για τα 2 εκατομμύρια από τον προπολογισμό και το ένα από τις χώρες μέλη. Και νομίζω ότι μέρος της συνεισφοράς του προπολογισμού πρέπει να γίνεται με αυτή την κατανομή. Αυτό είχα να πω. Και ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστούμε για αυτά που είπατε. Ο κύριος Σόλεκ, μέρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Στηρίζω τις επικρίσεις του όσον αφορά τις διαδικαστικές αδυναμίες που ανέφερε. Όμως έχουμε και κάποιες ανησυχίες για το πού πάνε τα χρήματα της διευκόλυνσης Είμαστε πολύ επικριτικοί για την σχέση αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Δεν μας αρέσει το γεγονός ότι έχουμε αναθέσει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά τη φύλαξη των συνόρων μας και θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα τι χρηματοδοτούν τα χρήματά μας. Ακούμε από διάφορες πηγές ότι αγοράστηκαν σκάφια από μια Ολλανδική εταιρεία με χρήματα από την τουρκική αυτή διευκόλυνση. Εγώ θέλω να ξέρω, να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχύει αυτό, ναι ή όχι. Και αν ισχύει, είναι συμβατό με την νομική βάση της διευκόλυνσης. Εμείς έχουμε κάποιες αμφιβολίες από αυτού. Νομίζουμε ότι το πεδίο δράσης της διευκόλυνσης δεν θα έπρεπε να πάει σε διαχείριση των συνόρων. Έχουμε και αμφιβολίες σε σχέση με το κατά πόσο τα χρήματα αυτά της διευκόλυνσης υπολογίζονται σαν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ή όχι. Γιατί νομίζω ότι αποδυναμώνεται έτσι η έννοια της αναπτυξιακής βοήθειας, δεδομένου μάλιστα που η Τουρκία δεν είναι αναπτυσσόμενη χώρα Και για μας οι κύριοι δικαιούχοι δεν είναι η Τουρκία. Υπάρχουν πολιτικά και οικονομικά ωφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, θα ήθελα αυτά τα δύο πράγματα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σολέ. Θα απαντήσει σε λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προηγουμένως η κυρία Κορταζαμπάλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, και εγώ σύντομα θέλω να στηρίξω την πρόταση του κυρίου Μουρεσάν με το διορθωτικό προϋπολογισμό αριθμός 3. Στηρίζουμε και εμείς την άποψη που είχε και ο συγητής του 2018 και του 2019 όσον αφορά ε, τα κονδύλια αυτά για την Τουρκία. Δεν είναι μόνο θέμα του να αφήσουμε κάποιο περιθώριο, να είμαστε προσεκτικοί για να μπορούμε να αντιδράσουμε, να έχουμε περιθώριο. Αυτό πάντα προσπαθούμε να το κάνουμε. Απλώ πάντα υπάρχουν τόσο πολλέ προτεραιότητε που φτάνουμε τον προπολογισμό στα οριά του. Εδώ όμω είναι θέμα συμπεριφορά του Συμβουλίου. Πώ παίρνει αποφάσει. Γιατί θυμίζω ότι ήμασταν σε διαπραγματεύσεις για ποιο προπολογισμό ήταν του 17 και μας έφτασε η πληροφορία ότι το Συμβούλιο είχε ήδη αποφασίσει. Οπότε είναι μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί. Και τώρα εμείς του προπολογισμού έπρεπε να φροντίσουμε να μας κάνει. Αυτό ήταν ε, το πρώτο κομμάτι της διευκόλυνσης για την Τουρκία. Τελικά βρήκαμε τα 2-3 ε, μάλλον αποφασίσαμε δύο το, το προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τις χώρες μέλη. Τώρα όμως τι θέλουνε. Θέλουν παραπάνω. Όμως πάντα το λέγαμε και στην περίπτωση της Τουρκίας ότι δεν είναι δυνατόν με κάθε ε, συμβούλιο, κάθε διάσκεψη κορυφής να μας το πετάνε το τραπέζι και εμεί να πρέπει να τα βολέψουμε και να αναγκαζόμαστε να πάρουμε χρήματα από το ένα για να τα βάλουμε στο άλλο. Δεν είναι σοβαρό. Ελπίζω στο επόμενο Συμβούλιο να ασχοληθούν σοβαρό όχι μόνο για ε, τα κονδύλια για την Τουρκία, γενικότερα με τη μετανάστευση, όπως και να έχει πάντως το πράγμα. Αυτή η πρώτη πρόταση διόρθωσης του 2018 πηγαίνει στη γραμμή των όσων έχουμε ζητήσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να υπάρξει καινούριο χρήμα, να μην κόψουμε απαλού. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με το δεύτερο σκέλος του προπολογισμού 2019. Θα ήταν σφάλμα πάντως να πάρουμε 1,5 για να χρηματοδοτήσουμε την διευκόλυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο να ζητάει το λόγο και εφόσον η Κομισιόν αντιπροσωπεύεται εδώ από τον κύριο Ιραέλα και τον κύριο Βανχεμ που είναι επικεφαλής για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία υπεύθυνο για το προενταξιακό μέσο Ποιος από τους δυο σας λοιπόν θα πάρει πρώτος το λόγο Κύριε Δουρέλα, μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με τη συμφωνία σας. Θα ξεκινήσω και μετά θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να συμπληρώσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Μουρισάν, τον Γενικό Εισηγητή για την επικοδομητική του προσέγγιση για αυτό το, για αυτό το θέμα και επίσης καταλαβαίνω ότι από τις παρεμβάσεις των σκιωδών ότι αυτή η προσέγγιση μάλλον υποστηρίζεται από όλους σας. Ήταν πολύ σημαντικό για μας την Κομισιόν να προχωρήσουμε σε μία ε, ε, προσέγγιση σε δύο βήματα. Πρώτον, επίγουσα ανάγκη να, χρησιμο... να ε, χρηματοδοτηθούν οι συμβάσεις των δασκάλων, 5.000 δάσκαλοι στην Τουρκία, που διδάσκουν περίπου 300.000 παιδιά των Συρίων προσφύγων. Είμαι πολύ χαρο... ευτυχής που αυτή η προτεραιότητα λήφθη υπόψη και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση σύντομα. Μπορώ επίσης να σας επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο έχει βρει ειδική πλειοψηφία για να προχωρήσει με το διευθυντικό όπως το πρότεινε η Κομισιόν ε, σήμερα, ε, μάλλον, συγγνώμη, αυτή την εβδομάδα αργότερα. Ε, τώρα, όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν από τον Σκιώδη των Πρασίνων, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μέσα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης έχουμε χορηγήσει 20 εκατομμύρια ευρώ υπό το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Για την εκπαίδευση της τουρκικής ακτοφυλακής ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε πλέον θύματα, προσφύγων, ε, θύματα πρόσφυγες που φεύγουν από την Τουρκία για τα νησιά. Μετά έχουμε ε, ε, ε, επίσης είναι αυτό επιλέξιμο. Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι επίσης επιλέξιμη υπό την χρήση αυτού του κονδύλιου. Όσον αφορά την Κομισιόν, αυτό το project αιτιολογείται και έχουμε διατηρήσει αυτή τη θέση στην αρμόδια ομάδα εργασία. Η ομάδα εργασία του ΟΣΑ το συζήτησε νωρίτερα φέτος και αποφάσισε ότι το 97% των χρημάτων του 2016 της διευκόλυσης ήταν ε, δυνατόν να ε, δαπανηθεί ε, το 2017. Εχθές είχαμε συνεδρίαση της Διευθυντικής Επιτροπής, Steering Committee, και αυτή υιοθέτησε το στρατηγικό σημειωμό ότι στο μέλλον όλα τα χρήματα που θα δαπανώνται από την διευκόλυνση ε, θα ε, μπαίνουν και στο προϋπολογισμό, θα μπαίνουν στο προσχέδιο, στο διορθωτικό με συγχωρείτε. Κύριε Γενικέ, εισηγητά, θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Νομίζω πως υπόθηκαν όλα και με σαφήνεια. Οπότε προχωρούμε προς μια συμφωνία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Δεν άκουσα κάποιον να διαφωνεί για την σύσταση του Γενικού Εισηγητή. Ο κύριος Σολέ ε, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση για τα πλοία. Μάλιστα. Να κλείσουμε τότε και να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Και τώρα διακόπτουμε, θα ξαναρχίσουμε σε 5 λεπτά με την ακρόαση που έχει προγραμματιστεί ώστε να δούμε πού βρίσκεται η πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των προσφύγων, ποια είναι η ανθρωπιστική δράση. Είχαμε μια πρώτη ακρόαση το Μάιο για, όσους, ε, για τα όσα γίνονταν εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα μιλήσουμε για τα κονδύλια που θα πανώνται εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Διακόπτεται η συνεδρίαση.